Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε. Ε, γιατί έχουμε αρκετά γεμάτη ημερησία διάταξη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής που εξετάζουμε την αναθεώρηση του κώδικα περιθεωρήσεων σήμερα, γιατί ήρθε σε επαφή μαζί μου ένας ε, μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος μου μίλησε για μια τεράστια κλίμακα διαφθορά ε, και μου περιέγραψε τι συμβαίνει. Ε, η Επιτροπή μας ε, έχει μια μακρά ιστορία ως φόρουμ, ως βήμα για πολλά θέματα μετανάστευσης, ηθαγένειας, ελέγχου των συνόρων. Ο χώρος Σέγγεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ένωση. Όλοι μπορούμε να ε, ταξιδεύουμε ε, χωρίς ε, πρόβλημα. Ωστόσο σήμερα και θέλω να θίξω ένα σοκαριστικό θέμα παράνομων θεωρήσεων και εμπορίου θεωρήσεων που έγινε και διαπιστώθηκε σε ένα από τα κράτη-μέλη μας. Κυκλοφορούν φήμες λοιπόν, ε, βάσιμες φήμες, ότι ένας υψηλά ιστάμενος ε, στην Μάλτα, αρμόδιος για την έκδοση θεωρήσεων, ε, παίρνει χρήματα για να εκδίδει τέτοιες θεωρήσεις στην Λιβύη. Μάλιστα φαίνεται ότι είναι αναμεμειγμένον και ο Μαλτέζος πρόξενος στην Τρίπολη. Η Καρίνση Γαλήσια φαίνεται φαίνεται πως είχε γράψει άρθρα το 13 ήδη όπου ισχυριζόταν ότι οι πρόξενοι της Μάλτας είχαν εκδώσει θεωρήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν δικαίωμα κανονικά. Οι τελευταίες εκθέσεις λένε πως η Μάλτα έχει εκδώσει 88.000 θεωρήσεις Σέγγεν, ε, συν αναρρύθμιτες ιατρικές θεωρήσεις ε, η Μάλτα έχει 400.000 ε, κατοίκους. Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Λιβύη, ο διακόπτη όμως ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, είπατε για διαδικαστικό. Ίσως θα ήταν καλό να είναι κομμάτι της συζήτηση σήμερα αυτό που λέτε για τον κώδικα περιθωρήσεων. Πόσο ακόμα θέλετε να μιλήσετε, έχετε ακόμα πολλά να μας πείτε, γιατί γιατί δεν είναι διαδικαστικό. Εντάξει, γενναιόδωρα σας άφησα να πάρετε το λόγο γιατί ε, ε, είστε τακτικό μέλος και είστε τακτικά παρόν. Νομίζω καταλάβαμε το θέμα σας, αλλά να το κλείσετε. Θέλω άλλο ένα λεπτό μου το δίνετε. Ναι, είμαι πολύ γενναιόδωρος σήμερα, αλλά παρακαλώ ένα λεπτό μόνο. Να έχετε τελειώσει ένα λεπτό. Um, η Λιβύη είναι ένα μέρος όπου χιλιάδες ε, θεωρήσεις Σέγγεν έχουν πουληθεί και ούτε ο Πρωθυπουργό ούτε η αστυνομία έχουν σωστά διερευνήσει το θέμα. Ακόμα και οι τοπικοί δημοσιογράφοι που ανέφεραν το θέμα ε, πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, ε, δίωξη, δικαστική δίωξη και να διωχθούν για απάτη. Όταν όμως η Δάφνη Καρουάνα Γαλήθια δολοφονήθηκε για αυτούς τους ισχυρισμούς, λόγω αυτών των ισχυρισμών της, νομίζω πως θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ πιο ε, εξονυχιστικά αυτή την υπόθεση. Όταν ερωτήθηκε ο Επίτροπο Αβραμόπουλο από την Ευρωβουλευτή Αναγκόμε σχετικά, απάντησε πω δεν ε, γίνονταν πωλήσει θεωρήσεων στη Λιβύη. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να ε, ερευνήσει αυτή τη θέμα, αυτό το θέμα και να το προσέξει, γιατί είναι μια φρικτή περίπτωση πώλησης θεωρήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ λέει Πρόεδρος. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Πρόεδρος της, της Νέας Ομάδας Εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα που ερευνά τέτοια ζητήματα είναι εδώ στην αίθουσα και θα πρότεινα λοιπόν να καταθέσετε γραπτή ερώτηση για αυτό το θέμα επίσης. Αλλά εμεί καταλάβαμε ακριβώς τι συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε. Και όπως σας είπα, σας έδωσα χρόνο γιατί τακτικά παρακολουθείτε και συμμετέχετε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Και τώρα να προχωρήσουμε. Α, συγγνώμη, ο κύριος Κοέλιο, διαδικαστικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω μόνο να σας πω σε εσά και στην Επιτροπή να σας ενημερώσω ότι ε, έγινε συζήτηση ε, στο θέμα της, για το θέμα της Μάλτας ε, στην ομάδα εργασίας για τον έλεγχο του Σέγγεν και συζητήθηκε ε, λόγω του ότι το ανέφερε η Άννα Γκόμες. Υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τη ε, του συστήματος θεωρήσεων από πλευρά μάλτα. Δεν θα επεκταθώ στα πορίσματα αυτά και στα στοιχεία που έχουμε. Πάντως έχουμε εγκύψει στο θέμα. Είναι ένα θέμα αρχής που κάποια στιγμή θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα της ισορροπίας ανάμεσα στις εθνικές αρμοδιότητες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Διότι η έκδοση θεώρηση είναι εθνική αρμοδιότητα και βεβαίως υπάρχουν κανόνες μέσα στο πλαίσιο το εθνικό. Όμως δεν έχουμε την ε, αρμοδιότητα να πούμε στα κράτη-μέλη όχι αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε. Και είναι επίσης ε, δυσκολότερο για την ε, ηθαγένεια. Είδαμε εκθέσεις, εκεί όπου αναφέρθηκε και ο συνάδελφος, είναι όλα αυτά πολύ ανησυχητικά, αλλά πρέπει να δούμε τι είδος τρόπους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φροντίσουμε αυτά τα θέματα που είναι ε, εθνικής αρμοδιότητας. Κύριε Σκρίπεκ, κοιτάξτε, δεν θέλω να ξεκινήσουμε συζήτηση, αλλά νομίζω ο Κοέλιο προσπαθεί εδώ να βοηθήσει. Δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει κάποιο... Ε, υπάρχει εδώ βάσιμε, ε, ε, ε βάσιμα το θέμα, υπάρχουν στοιχεία και υπάρχουν συνάδελφοι που γνωρίζουν επίσης ότι συμβαίνει αυτό. Καλά κάνατε που παρενέβητε, αν και δεν ήταν ε, στην ημερήσια διάταξη. Ωραία, λοιπόν, τώρα περνάμε στο πρώτη, στην πρώτη συζήτηση που είναι η παρουσίαση από την πλευρά της Επιτροπής του νέου κώδικα θεωρήσεων. Ο Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγιγιάρ είναι ο δικός μας εισηγητής και ο κώδικας θεωρήσεων ορίζει τις διαδικασίες και τους όρους για την έκδοση θεωρήσεων για στόχους σύντομης διαμονής ή ε, διέλευσης. Ε, είναι σκόπιμο να διευκρινίζονται αυτές οι συνθήκες και να βελτιώνονται τα διαδικαστικά ε, δικαιώματα. Δεν έχει αναθεωρηθεί από το 2010 και το 2014 η Κομισιόν υιοθέτησε μία προτινόμενη ε, αναθεώρηση, όμως λόγω αποκλήσεων ε, στις θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις παρά τις σημαντικές προσπάθειες και την επιμονή της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου και η ε, σημερινή παρουσίαση θα συμπληρωθεί από παρουσίαση και ανακοίνωση της Επιτροπής όπου προσαρμόζεται κοινή προεπτική ε, θεωρήσεων στις νέες προκλήσεις. Πρώτα θα δώσω το λόγο λοιπόν στον, εκπρόσωπο της Επιτροπής και μετά στον εισηγητή μας Χουάν Φερνάντο Λόπεθ Αγγιλάρ ε, και στους κοιόδης στη συνέχεια ή όποιους άλλους συναδέλφους θέλουν να το λόγο. Θα ζητήσω λοιπόν πρώτα από την Επιτροπή να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Yes, good morning. Thank you, Mr. Καλημέρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Όντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Μαρτίου υπέβαλε ανακοίνωση για το πώς θα πρέπει να προσαρμοστεί η πολιτική θεωρήσεων στις νέες προκλήσεις. Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2017 πάνω από 16 εκατομμύρια για σύντομη διαμονή. Άρα η πολιτική θεωρήσεων πρέπει να είναι τέτοια που να διευκολύνει τους επισκέπτες να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο ευνοεί την ευρωπαϊκή οικονομία. Έτσι. Ε, ενισχύεται κατά 10% το ευρωπαϊκό ΕΠ. Συγχρόνως ε, βέβαια αντιμετωπίζουμε και άλλες προκλήσεις μεταναστευτικού τύπου, άρα πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική μας θεωρήσεων ανάλογα. Και η Επιτροπή θέλει να προχωρήσει, να υπάρχει συνοχή όσον αφορά την πολιτική μας θεωρήσεων, να δούμε τις εξωτερικές μας σχέσεις, να υπάρχει συνοχή επίσης με άλλες πολιτικές μας. Ο ειδικό μηχανισμός που προβλέπεται από τον κανονισμό 39 που αναθεωρήθηκε πέρυσι προσθέτει και άλλο ένα στοιχείο και υπάρχουν συγχρόνως και εξελίξεις στα συστήματα ενημέρωσης όπως το σύστημα εισόδων-εξόδων, το αιτίας, ε, διαλειτουργικότητας κλπ. Όλες αυτές οι εξελίξεις συνεισφέρουν προκειμένου να μειωθεί η παράτυπη μετανάστευση και η κινδύνη στην, και η στην ασφάλεια. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε άλλη πρόταση στο παράρτημα 2 αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν βάσει ακριβώς ε, αυτών. Για να είμαστε τώρα πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων για θεώρηση και να ενισχυθούν οι έλεγχοι για την ασφάλεια και να αποφύγουμε να επιτρέψουμε την είσοδο σε ανθρώπους που απειλούν απειλή, στις 16 Μαΐου ζητήσαμε το σύστημα SIS να αναβαθμιστεί Όσον αφορά το μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ξεκινήσει συζήτηση για την παρατέρω ψηφιοποίηση τη προσέγγιση αυτή. Να χρησιμοποιούνται δηλαδή νέε τεχνολογίε για να διευκολυνθεί η επεξεργασία των δεδομένων προ όφελο των χωρών μελών αλλά και των ανθρώπων που υποβάλλουν αιτήσει για θεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τι τροπολογίε. Απέσυρε την πρότασή τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναδιατύπωση. Υπάρχει, υπήρχε μια πρόταση για την αναθεώρηση το Μάρτιο μαζί με την ανακοίνωσή μας και η πρόταση αυτή έχει σαν στόχο η κατάσταση να γίνει περισσότερο ασφαλής όσον αφορά την επεξεργασία των αιτήσεων. Ε, σας είπα, άλλαξα η κατάσταση ασφάλειας εξαιτίας του μεταναστευτικού Εξού και υπήρχε η πρόταση αναδιατύπωση του 2014. Η πρόταση πάντω περιλαμβάνει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται τελικά στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναδιατύπωση, που έχουν να κάνουν με την απλοποίηση τη διαδικασία. Η Επιτροπή, για παράδειγμα, πρότεινε να μπορεί κανεί πολύ νωρίτερα να υποβάλει αίτηση για θεώρηση πολύ νωρίτερα από ό,τι έχουν σχεδιάσει τα ταξίδια τους οι πολίτες ώστε να υπάρχει πιο έγκαιρα και απάντηση και οι προθεσμίες να είναι πιο μικρές που έχουν δηλαδή τα προξενία στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν αν θα χορηγήσουν τη θεώρηση ή όχι. Επίσης για τα μικρά τουριστικά ταξίδια να μπορεί κανείς να εστίσει στη θεώρηση στα εξωτερικά σύνορα. Να υπάρχουν κάτι προσωρινά προγράμματα δηλαδή γι' αυτό να μπορεί να γίνει φυσικά καλός έλεγχος των στοιχείων του ετούντος και συγχρόνως όσοι ταξιδεύουν τακτικά να μπορούν να αποφεληθούν από ένα άλλο σύστημα, δηλαδή να μην περνάνε κάθε φορά από την ίδια βαριά διαδικασία κάθε φορά που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να υπάρχει και μια θεώρηση για πολλαπλές εισόδους. Μια άλλη αλλαγή που προτείνεται στην πρόταση είναι η επεξεργασία των αιτήσεων για θεωρήσει που είναι όλο και περισσότερες κάθε χρόνο να γίνονται πιο απλοποιημένα. Τα τέλη παραμένουν ίδια από το 2006 και λέμε τώρα από 6 να πάνε στα 8 ευρώ. Είναι μια μικρή αύξηση που λαμβάνει υπόψη Εξάλλου είναι λιγότερο αυτό που ζητάμε εμείς από ό,τι ζητάνε άλλες χώρες να έχετε υπόψη σας, έτσι. Αλλά Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και με τα ποσά αυτά οι χώρες μέλη θα μπορούν να διατηρήσουν το προσωπικό που χρειάζονται τα προξενία για να επεξεργάζονται τις αιτήσει για θεωρήσεις και θα μπορεί έτσι να γίνεται καλός έλεγχος. Τέλος, η πρόταση θέλει να διασφαλίσει ότι η κοινή μας πολιτική για θεωρήσεις θα βελτιώσει και τις ε, σχέσεις μας με τρίτες χώρες όταν πρόκειται για την επιστροφή, την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών. Θέλουμε πιο αυστηρές προδιαγραφές για την επεξεργασία ε, των θεωρήσεων, άπαξ και η τρίτη χώρα δεν είναι συνεργάσιμη, να υπάρχει και η εξέταση κατά περίπτωση, αξιολόγηση και να λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια. Είναι σαφές ότι αυτή η νέα προσέγγιση δεν έχει επιπτώσεις στα δικαιώματα των ετούντων θεώρηση. Μπορούν πάντα, εξίσου όπως και παλιά, να υποβάλουν αίτηση και να παίρνουν απάντηση μετά από την κατάλληλη επεξεργασία. Η Ευρώπη θέλει να είναι στον τουρισμό, στους επιχειρηματίες, στους ταξιδιώτες γενικά, αυτούς που επισκέπτονται τις οικογένειές τους, αλλά συγχρόνως προσαρμόζουμε τους κανόνες μας για να ε, τους προσαρμόσουμε στις νέες καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε ότι είμαι στη διάθεση των μελών της Επιτροπής σας, του εισηγητού, των σχεδόν εισηγητών, για να προχωρήσουμε. Ωραία, τώρα το λόγο έχει ο εισηγητής ο κύριος Λόπες Άγγιλαρ. Εκτός μικροφώνου. Με συγχωρείτε. Προσπαθώ να παρουσιάσω το θέμα δεδομένου ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε γι' αυτό. Όπως γνωρίζετε έχει περάσει αρκετός καιρός ε, κατά τον οποίο συζητούμε αυτό το θέμα και με τους κοιώδεις εισηγητές. Η συνεργασία μας είναι πολύ στενή και γόνιμη. Όμως υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα και έχουμε απόλυτη επίγνωση του ότι πλησιάζει το τέλος της θητείας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επομένως πρέπει η δουλειά να έχει ολοκληρωθεί ε, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Προσπαθώ λοιπόν να σας παρουσιάσω την κατάσταση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή για την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός κοινού ε, κώδικα για τις θεωρήσεις. Ο κώδικας για τις θεωρήσεις, όπως γνωρίζετε, είναι ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής θεωρήσεων και η νομική βάση είναι η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν νομική βάση έτσι ώστε το Κοινοβουλίο να νομοθετήσει για μια νέα πολιτική και νέα νομοθεσία για τις θεωρήσεις, για να επέλθει μια εναρμονισμένη διαδικασία για την επεξεργασία αιτήσεων ε, θεώρησης και την έκδοση θεωρήσεων για ε, ε σύντομες και ε, διελεύσεις ε, αεροδρόμια μέχρι 90 ημέρες. Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν έχει αναθεωρηθεί από το 2010 όποτε και σε ισχύ. Και το αρχικό σκεπτικό ήταν ε, η διευκόλυνση και το να αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση αυτή δεν είναι η πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τον Απρίλιο του 2014 για πρώτη φορά μία πρόταση αναθεωρ... αναδιατύπωσης του κώδικα για τις θεωρήσεις και μετά είχαμε προβλήματα με τη θέση του Συμβουλίου. Οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν παραπέρα παρά τις ε, προσπάθειες που καταβάλαμε και παρά την ε, δουλειά όλων των ε, συναδέλφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αντίθετη στην ε, εισαγωγή μιας ανθρωπιστικής θεώρησης στον κώδικα αυτό. Ήταν κάτι το οποίο ζητούσαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι συμμετέχοντες διαπραγματεύσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, συμβούλια, όλοι ζητούσαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχει μία νόμιμη οδό άφηξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε οι έχοντες ανάγκη να μπορούν να αιτηθούν ανθρωπιστικής προστασίας. Το Συμβούλιο όμως αρνήθηκε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για ε, το θέμα αυτό εάν δεν αποσύρονταν οι τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν μας πήρε δύο χρόνια μέχρι να βρούμε μια συμβαστική λύση και τότε μας ζητήθηκε να αποσύρουμε τις ε, τροπολογίες μας. Όπως γνωρίζετε ζητήσαμε να εκδώσουμε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη δική της πρόταση για τον ε, κώδικα των θεωρήσεων. Δυστυχώς όμως το Συμβούλιο συνεχίζει να μπλοκάρει τις ε, εξελίξεις παρά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής σκοπεύει στο να διευκολύνει τους, τους καλόπιστους ταξιδιώτες ταυτόχρονα εγγυόμενη την ε, ομαλή λειτουργία του συστήματος. Στο, στο πλαίσιο λοιπόν της ε, μετανάστευσης είναι πολύ σημαντικό οι θεωρήσεις να εξεταστούν μαζί με τους ελέγχους στα σύνορα. Το Συμβούλιο βέβαια έχει κάποιες αιμονές θα λέγαμε με τους ελέγχους και την ασφάλεια στα σύνορα και το 2018, φέτος δηλαδή, πρόκειται να, υπάρχουν εξελίξ, να υπάρξουν εξελίξεις για το σύστημα VIS. Θα ληφθούν λοιπόν αποφάσεις σχετικά με την εξέταση των αιτήσεων, με τα τέλη, με τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν, με την ιατρική ασφάλιση και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα τεχνικά οι τεχνικές αυτές λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι καλόπιστοι ταξιδιώτες να ταξιδεύουν εντό Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς προβλήματα. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η αναδιατύπωση της ε, νομοθεσίας για πολλού τομεί και για τις επιχειρήσεις και για τον τουρισμό και για σπουδές, για έρευνα. Ε, για θέματα δηλαδή ουσιαστικά και πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει λοιπόν η Ένωση να εργαστεί προς επιτεύξη αποτελεσμάτων και ε, να εξισορροπήσει τις ε, ανησυχίες για το μεταναστευτικό με τις πρακτικές δυσκολίες του θέματος. Για μένα προσωπικά οι ανησυχίες αυτές για τη μετανάστευση έχουν άμεση σχέση με τον κώδικα για τις θεωρήσεις, αλλά πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα. Υπάρχει και θέμα προσωπικών ε, δεδομένων, γι' αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί και ο επόπτης προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν θέματα ασφαλείας, σίγουρα, όμως ε, τα ζητήματα ασφαλείας και καταπολέμηση δημοκρατίας κάπως... Ε, δεν αφήνουν περιθώριο για να δούμε την ουσία και νομίζω πως ε, στην παρούσα πρόταση δεν θα έπρεπε να επισκιάζουν τις ε, διαπραγματεύσεις, διότι μην ξεχνάμε εδώ πρόκειται για καλόπιστους ε, ταξιδιώτες, για τη χορήγηση θεωρήσεων σε αυτούς. Και θα έλεγα ότι πραγματικά επισκιάζουν τις, ε, οικονομικές, τους ε, ταξιδιώτες που ταξιδεύουν για οικονομικούς ε, ή άλλους σκοπούς. Όμως, το βυφιστάμενο πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο στο οποίο συμμετέχει και, ε, το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο συνομοθέτης. Έχουμε το άρθρο 25α, ε, το οποίο περιγράφει την υποχρέωση συνεργασίας για την πολιτική εισόδου, επανεισόδου. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο έχουν προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ποτέ μέχρι τώρα, μέχρι τώρα όμως δεν έχει φτάσει σε ε, σημείο να συμπεριληφθεί σε μια νομοθετική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μπορεί να συνεισφέρει στην επανιστοχή των ε, νόμιμων ε, μεταναστών και των ταξιδιωτών για επαγγελματικούς σκοπούς. Όπως ε, είπα και πριν, το αρχικό σκεπτικό ήταν τελείως διαφορετικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα μέτρα για τις θεωρήσεις δεν αρκούν από μόνα τους για να αλλάξουν το σύστημα χορηγήσης θεωρήσεων. Χρειάζεται πολιτική βούληση και συνεργασία σε πάρα πολλούς τομείς, στο εμπόριο, στην ε, εκπαίδευση έτσι ώστε να συνεργαστούν ε, όλες οι τρίτες χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, γίνεται λόγος για έλλειψη ε, στοιχείων. Είμαι σύμφωνος με αυτό. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να δούμε πώς, μπορού, πώς μπορεί αυτή η νέα πρόταση να οδηγήσει στην διευκόλυνση ε, των, ε, της χορήγησης ε, θεωρήσεων, στη βελτίωση της κατάστασης. Βέβαια, μας έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η παρούσα νομοθεσία δεν έχει χώρο για συζήτηση περί ανθρωπιστικής βοήθειας και λοιπόν θεμάτων, όμως δεν το θεωρούν και απίθανο να γίνει ο κώδικας θεωρήσεων ένα εργαλείο για ε, την επαναπροώθηση μεταναστών. Να του στέλνουν πίσω από εκεί που ήρθαν δηλαδή με λίγα λόγια. Η εκτίμηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζει ε, τα στοιχεία αυτά ε, αναφέρεται στην αύξηση της μόχλευσης για τις μη συνεργαζόμενες χώρες, αυξάνει τις ε, απαιτήσει σύμφωνα με τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη νομοθεσία. Όμως, πιστέψτε με, ως εισηγητής της έκθεσης αυτής και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους και εισηγητές θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μας θα εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά έτσι ώστε να περάσουμε αυτή την νομοθεσία και να την κάνουμε πραγματικότητα, να ολοκληρωθεί το νομοθετικό μας έργο πριν το τέλος της ε, θητείας αυτής. Θεωρώ επίσης λυπηρό το γεγονός ότι έχουμε φτωχά αποτελέσματα στο θέμα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία μπλοκάρονται στο Συμβούλιο. Δεν μας ικανοποιεί καθόλου αυτό, διότι οδεύουμε προς το τέλος της θητείας μας και πραγματικά είναι πενιχρά τα αποτελέσματα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να εγκριθεί επιτέλους η νομοθεσία. Εμείς νομίζω πως κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε και Φυσικά προσπαθούμε να προτείνουμε ε, τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής έτσι ώστε να γίνει κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα περάσω τώρα αμέσω ε, στους κοιόδες ηγητές, αρχίζοντας με τον κύριο Μπέκερ εκ μέρους του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον ε, κύριο εισηγητή για την παρουσίασή τους. Συμφωνώ μαζί σας 100% η δουλειά που έχουμε κάνει είναι εξαιρετική και χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία νομίζω πως εστιάζει στα ουσιώδη, στις ε, ουσιώδεις αλλαγές και απαιτήσει έτσι ώστε στο μέλλον ε, να βελτιωθεί σημαντικά η νομοθεσία αυτή. Και ε, χαιρετίζω επίσης την ανθρωπιστική διάσταση με την ανθρωπιστική, χωρίς ανθρωπιστικής θεώρησης, διότι επιτέλους έπρεπε να συζητηθεί το θέμα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, σύνδεση με τα θέματα ασφαλείας, νομίζω πως η συζήτηση αυτή στην ε, παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει εξαντληθεί θα έλεγα. Γι' αυτό ελπίζω η ψηφιοποίηση, η πλήρης μάλιστα ψηφιοποίηση της ε, διαδικασίας χορήγησης και έκδοσης θεωρήσεων να είναι ε, κάτι που θα γίνει πραγματικότητα, όπως μας έχει ανακοινώσει η Επιτροπή. Σίγουρα δεν έχουμε ακούσει την τελευταία τους ε, λέξη, όμως ε, θεωρώ ότι το βασικό σκεπτικό, δηλαδή οι αθλητές, οι τουρίστες, οι ομάδες ε, ταξιδιωτών, οι επαγγελματίες, όλες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την δυνατότητα να ε, λαμβάνουν ε, θεώρηση βρεχίας διαρκείας με πολύ σύντομες και απλές διαδικασίες. Ελπίζω το θέμα αυτό να χειριστεί με τη δέουσα σοβαρότητα. Αυτό που χαιρετίζω επίσης είναι το ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι απόλυτα ανταγωνιστική όσον αφορά το κόστος. Η απλούστευση της όλης διαδικασίας είναι αποφασιστική σημασίας, ε, πιστεύω, διότι ακριβώς δίνεται έμφαση στους καλόπιστους ταξιδιώτες και ανταμείβονται οι ταξιδιώτες αυτοί ακριβώς για την καλή τους πίστη με την ε, επίσπευση της ε, διαδικασίας. Γι' αυτό έχουμε προτείνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή να λάβει χώρα στις 5 Νοεμβρίου, νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία και θα χαρώ πάρα πολύ αν αυτό γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. ευχαριστούμε πολύ. ECR. αντικαθιστάτε την κυρία Στίβενς, νομίζω που είναι σκιώδη, σωστά. Κύριε όχι, α, τότε αργότερα θα πάρετε εσείς το λόγο. Ο κύριος Ντεπρέ, σκιώδης από την ομάδα των φιλελεύθερων. Άλντε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, κάποια φιλικά λόγια προς τον εισηγητή Λόπες Αγγιλάρα. Γι' αυτόν και τους σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες ομάδες Εγώ θα παρουσιάσω τη θέση της ομάδας μου και δεν δεσμεύομαι από την ερμηνεία που δίνει στην θέση μας ο κύριος Λόπες Αγγιλάρη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πιστεύω ότι αποτελεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να βοηθήσουμε τους καλόπιστους ταξιδιώτες να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και από την άλλη διατηρώντας το στοιχείο της ασφάλειας με τους ελέγχους στα σύνορα. Τώρα, στην τωρινή πρόταση τη επιτροπή υπάρχουν κάποιες αλλαγέ σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση πριν από τέσσερα χρόνια. Για διάφορα σημεία και σημαντικά. Που δεν αιτιολογούνται όμως. Τι σας έκανε να αλλάξετε τόσο πολύ διάφορα σημεία σε σχέση με την πρόταση που είχαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Δεν το καταλαβαίνω τι καταστροφή προβλέπετε όσον αφορά το ανθρωπιστικό. Συζητήσαμε πολύ με την προηγούμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τους Κιώδης, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τίποτα δεν προχωράει αν συνεχίζουμε να απαιτούμε η ανθρωπιστική βίζα να συμπεριλαμβάνεται στον κώδικα για τις θωρήσεις. Τώρα δεν θέλω να ξαναρχίσω εδώ το τσίρκο που είχαμε και την προηγούμενη φορά που τσακώθηκαμε και δεν καταλήξαμε πουθενά. Τώρα συζητάμε τον κώδικα για τις θεωρήσεις. Τώρα για τις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας. Εδώ βλέπω τρεις κατηγορίες εγώ. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν τα πράγματα με τα οποία συμφωνούμε. Ακόμα και αν έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Πρώτον, πιστεύουμε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια μικρή αύξηση του κόστους των θεωρήσεων, δεδομένου ακριβώς ότι έχουμε πολύ περισσότερες αιτήσει. Βέβαια όταν βλέπω ότι για τα παιδιά 6 έως 12 ετών πάμε από τα 5 στα 40 ευρώ, ε, για εξηγήστε το μου αυτό, πώς γίνεται σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση. Έπειτα, χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι οι αιτήσει θα μπορούν 6 μήνες πριν να υποβάλλονται, οι αιτήσει δηλαδή αντί για 3, ότι θα είναι πιο σύντομο το διάστημα προκειμένου να ξέρει ο ετών την απόφαση και εγώ θα πήγαινα πιο μακριά και θα έλεγα γιατί να μην πάμε στις πέντε μέρες όταν υπάρχουν βιομετρικά στοιχεία ήδη. Δεν βλέπω γιατί να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και να περιμένουμε δέκα μέρες ενώ υπάρχουν τα βιομετρικά δεδομένα, ό,τι χρειάζεται δηλαδή κανείς για να αποφασίσει. Και επίση μα χαροποιεί ιδιαίτερα η θέληση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, παρά τι επιφυλάξει του Συμβουλίου, να εισάγει την πρόταση της θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων. Πιστεύω ότι είναι κάτι καινοτόμο στην πρόταση και καλό. Τώρα, η δεύτερη κατηγορία είναι η... τα στοιχεία αυτά στην πρόταση για τα οποία έχω κάποιες επιφυλάξεις. Προβλέπεται προσφυγή όσον αφορά τους εξωτερικούς παρόχους. Αντί να είναι δηλαδή το προξενείο, να υπάρχει δυνατότητα να έχουμε κάποιους εξωτερικούς παρόχους. Εδώ, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας φιλελεύθερος που όμως ακολουθεί κανόνες. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα οι κρατικές αρχές να έχουν την ε, ευθύνη. Οπότε αναρωτιέμαι επί της αρχής, αλλά και για το τεχνικό σκέλος. Δηλαδή, καταλαβαίνω καλά, δηλαδή αναθέτουμε στον εξωτερικό πάροχο το καθήκον να πάρει αυτός δακτυλικά αποτυπώματα και βιομετρικά χαρακτηριστικά. Σωστά, το καταλαβαίνω. Ε, ωραία, τότε ένα λόγο παραπάνω να κάνω την ερώτησή μου επί της αρχής. Οπότε, επαναλαμβάνω, έχουμε επιφυλάξεις για την αύξηση της τιμής όσον αφορά τα παιδιά και για τη σχέση της ε, θεώρησης με τους εξωτερικούς παρόχους. Είμαι φιλελεύθερος, αλλά με αυτό έχω πρόβλημα. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι είναι μια μικρή λεπτομέρεια για τι συμφωνίες που κάνουμε με άλλες χώρες. Αλλά εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπάρχει μείωση για του υπηκόους των χωρών που έχουν δεχτεί την επανεισδοχή. Ενώ εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει το κόστος. Δηλαδή τελικά θα είναι οι πολίτες αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν την ε, διάθεση της χώρας να κάνει να μην κάνει συμφωνίες επανεισδοχής. Και έρχομαι και στο τελευταίο, όπου θέλω περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαβάζω την πρότασή σας, αλλά δεν βλέπω τη δυνατότητα εισαγωγής ψηφιακής θεώρησης διάβασα. Μιλάτε για βινιέτ. Μα είμαστε στην ψηφιακή εποχή. Θα μπορούσαμε αντί να στέλνουμε αυτό το χαρτάκι με ό,τι επιπλέον κόστος ή και προβλήματα ασφάλειας και προκύπτει, θα μπορούσαμε να το στέλνουμε ηλεκτρονικά. Μα έτσι κι είναι στο SIS όλες οι θεωρήσεις, έτσι δεν είναι. Οπότε γιατί πρέπει να είναι και σε χαρτί. Θα ήθελα λοιπόν παρακαλώ να μου απαντήσετε για ποιο λόγο δεν έχετε προβλέψει την ψηφιακή θεώρηση. Κατά τα άλλα θα συμμετάσχει ενεργά η ομάδα μου στις συζητήσεις που θα γίνουν προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον νέο κώδικα θεωρήσεων και να καταφέρουμε να έχουμε και μια ανθρωπιστική θεώρηση βίζα σε διαφορετικό όμως φάκελο, χωριστά. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει στο τέλος βέβαια. Αλλά προηγουμένως η κυρία Βαλέρο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα έχω ξαναπεί αυτά και στο παρελθόν. Μπορώ να συμφωνήσω με την περιγραφή του πλαισίου και όντως πιστεύω και εγώ ότι έχουμε μια καλή πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκρίνοντας, αν μη τι άλλο, με την αρχή αυτής της θητείας. Εμένα όμως στη θέση μου ότι οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις είναι κάτι καλό και είναι κάτι που θα μπορούσε και θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόταση. Θα ήταν απόλυτα φυσιολογικό να συμπεριληφθεί εδώ. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν θα τα καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό αυτή τη φορά. Είναι σαφές. Θα ήταν όμως ε, το καλύτερο μέρος να συμπεριλάβουμε την ανθρωπιστική θεώρηση. Τώρα, αν ε, εξετάσουμε την ε, πρόταση αυτή που έχουμε μπροστά μας σήμερα, είναι κρίμα που θέλουμε να διευκολύνουμε τα πράγματα για τους τουρίστες, τους φοιτητές, τους επισκέπτες, όλο τον κόσμο. Έτσι αυτή ήταν η ιδέα. Να είναι πιο εύκολο να έρχονται στην Ευρώπη οι επισκέπτες. Ενώ έχουμε μπροστά μας μία πρόταση που έχει αλλάξει στόχο από ό,τι βλέπω και λέει να γίνει πιο αυστηρή η πολιτική θεωρήσεων, ώστε να αποτελέσει ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση της ε, μετανάστευσης και άλλων αντίστοιχων προκλήσεων. Μα αυτή είναι μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που είχαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Αυτό αποτελεί μια τεράστια αλλαγή για μένα στην πρόταση. Συνεπώς είμαι κατά της αλλαγής αυτής. Εννοείται ότι θέλουμε ακόμα οι τουρίστες να έρχονται εύκολα στην Ευρώπη. Αν όμως συγχρόνως αυξάνουμε το κόστος από 60 στα 80 ευρώ και 35 με 40 για τα παιδιά και ξέρετε οι οικογένειες συχνά ταξιδεύουν με τα παιδιά τους οπότε για βάλτε τα όλα αυτά μαζί Έπειτα είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται πάρα πολύ στο χαρτί. Οπότε για να καταφέρει να συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα που χρειάζεται κανείς για να ταξιδέψει είναι δύσκολο. Τρομάζει ο κόσμος έτσι. Και αν απορριφθεί η αίτηση θεώρησης, ε, κάνεις τη θεώρηση για να πας και να υιοθετήσει, ας πούμε, δύο παιδιά. Και τελικά απορρίπτεται η θεώρησή σου. Τι γίνεται, σου δίνουν πίσω τα χρήματα θα έπρεπε να προβλέπετε κάτι τέτοιο. Να λέει δηλαδή μια διάταξη ότι αν υπάρξει απόρριψη τα χρήματα θα επιστραφούν. Θα ήταν πολύ καλό αυτό. Έπειτα στο άρθρο 25 μιλάμε για τη συνεργασία όσον αφορά την επανεισδοχή, τις επιστροφές. Εδώ δυσκολεύομαι να καταλάβω ποιος καλύπτεται από αυτή τη διάταξη. ιδίω το 5 θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου εξηγήσει ακριβώς ποιον εννοεί. Ποιος είναι αυτός που θα τύχει επανεισδοχής. Όλοι οι πολίτες, κάποιες κατηγορίες πολιτών. Μου φαίνεται σαφής η διατύπωση. Έπειτα υπάρχει το δίκτυο, η οργάνωση για, που είναι ιδιωτική για τον τουρισμό στην Ευρώπη, που είναι ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στην πρόταση αυτή. Κυρίως όσον αφορά την αύξηση του κόστους. Μας έστειλαν τη γνωμοδότησή τους και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να λάβουμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις τους. Η βασική ιδέα εδώ θα έπρεπε να είναι η απλοποίηση, να είναι πιο εύκολο να έρθει κανείς στην Ευρώπη και όχι να τους δυσκολέψουμε τη ζωή και να τους ξαναστέλουμε πίσω. σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Κοέγιο είναι ακόμα μιλητής. Κάνες άλλος. Και εσείς κύριε Σκρίπλετ είπατε ότι θέλετε να μιλήσετε στο τέλος, ε. Ναι, ναι, ακούω και εγώ τους συναδέρφους. Τους άκουσα. Άκουσα και τον κύριο Λόπες Αγγιλάρ. Είπατε ότι υπάρχουν εκατομμύρια ταξιδιώτες καλόπιστοι. Ναι, αλλά εδώ βάζουμε σε κίνδυνο τους Ευρωπαίους πολίτες. Μιλάμε για τη θεώρηση, για τις θεωρήσεις Σέγγεν, αλλά η Επιτροπή μας θα έπρεπε να ερευνήσει πόσες τέτοιες θεωρήσεις Σέγγεν ή για ιατρικούς λόγους δίνονται καταχρηστικά. Και το θέμα της εξωτερικής υπηρεσίας που θα μπορούσε να παίρνει τα δακτυλικά αποτυπώματα, το βρίσκω τρομερό αυτό, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε διαφθορά και να υπάρχουν και κενά να κλαπούν θεωρήσεις. Κύριε Κοέγιο, εσεί είπατε ότι είναι εθνική αρμοδιότητα αυτή η τραγική περίπτωση στη Μάλτα. Ναι, αλλά εμείς μπαίνουμε σε κίνδυνο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε απλώς ότι είναι εθνική αρμοδιότητα. Ο έλεγχο είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Θα έπρεπε να γίνεται έλεγχο. Τώρα υπάρχουν χιλιάδε θεωρήσει που έχουν απολυθεί. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό πάνε στη Λιβύη, δηλαδή οι μαχητές του ISIS ταξιδεύουν ελεύθερα και από την Λιβύη έρχονται σε εμά. Πόσοι φωτομεταλλιστές δεν υπάρχουν εδώ σε διάφορα κέντρα και κοιμούνται στα μέρη μας. Τι άλλο θέλουμε. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ αυτούς τους φοβερούς ισχυρισμούς. Πριν από δύο μέρες η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια της Μάλτας για να ερευνηθεί. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε όλη αυτή την υπόθεση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε σε κάποιον άλλον την υπόθεση αυτή. Αν θέλουμε ε, ανθρωπιστική ή άλλη θεώρηση, θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος και στην περίπτωση της Μάλτας. Δώστε προσοχή σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ο κύριος Σκόγιο και η κυρία Σίπελ και μετά θα επιστρέψουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πάρει το λόγο και ο συγκεκριτής ο κύριος Λόπες Άγγελαρ φυσικά. Ναι, ένα λεπτό μόνο. Και αυτά που λέει ο κύριος Σκρίπελ, εγώ δεν είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι όντως ανησυχητικά αυτά που διαβάζουμε στον τύπο. Ειλικρινά, όλες οι πληροφορίες είναι ανησυχητικές. Όμως, το πιο προβληματικό και από τις θεωρήσεις είναι η πώληση της υπηκότητας. Αν η Μάλτα πουλάει την ε, υπηκότητα σε κάποιους, ουσιαστικά πουλάει και την ευρωπαϊκή θαγένεια. Συνεπώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, αλλά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί το μεγαλύτερο μέρο της αρμοδιότητας είναι εθνική. Συνεπώς να είμαστε προσεκτικοί για το τι θα κάνουμε. Ποτέ όμως δεν είπα ότι πρέπει να το ξεχάσουμε και δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Είναι ανησυχητικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έρχομαι τώρα στο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Έχω ένα σύντομο σχόλιο για τον κώδικα θεωρήσεων. Η πρόταση αυτή είναι πράγματι σημαντική. Κυρίω αν δούμε το γενικότερο πλαίσιο που είναι καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών μα συνόρων. Έχει σημασία η νομοθεσία αυτή και αυτό φαίνεται και από τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει μέσω του τουρισμού. Συνεπώς αυτό θα ήθελα να το τονίσω ως εισηγητής για τις θεωρήσεις και θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις. Η πρόταση για τροποποίηση του συστήματος SIS δεν μπορεί να γίνει χωρίς κώδικα θεωρήσεων. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους βέβαια δεν μπορεί επίσης να χωριστεί το θέμα αυτό και από την διαλειτουργικότητα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν εξαιρέσει, βέβαια, που απαιτούν ταχεία δράση. Όμως, ως Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η θέση μας είναι συνεκτική. Προσφέρει συνοχή για ό,τι γίνεται στα εξωτερικά σύνορα. Είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ με όλους τους κοιόδες εισηγητές για όλα αυτά τα συναφή ζητήματα και φυσικά και για τον κώδικα θεωρήσεων. Και τώρα, παρακαλώ, κύριε Σίπελ. Ναι, σύντομα κι εγώ, γιατί λέμε και ξαναλέμε για τον έλεγχο των συνόρων μας εξαιτία του Ισλαμιστικού ε, της ε, Ισλαμιστικής ε, απειλής και τρομοκρατίας. Χτες συναντηθήκαμε με τον εκπρόσωπο της Europol που είπε ότι οι περισσότερες επιθέσεις που έχουν γίνει ή απόπειρες επιθέσεων που έχουν γίνει είχαν να κάνουν με αποσχιστικές τάσεις, με εθνικισμούς με ε, δεξιά και αριστερή ε, ακραία αντιμετώπιση. Οπότε αυτό να το έχουμε υπόψη μας όταν προσπαθούμε να πάρουμε τα σωστά μέτρα, έτσι. Πρόεδρος, ωραία. Καταλάβαμε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ να απαντήσει σε αυτά που είπε ο κύριος Ντεπρέ αλλά και οι υπόλοιποι, έτσι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, θα προσπαθήσω όντω να απαντήσω σύντομα. Για τη σχέση της πολιτικής θεωρήσεων και την επανεισδοχή. Είπα ότι είναι ένα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία των χωρών επανεισδοχής. Δεν λέω ότι είναι το μόνο, είναι και άλλα θέματα, ανάπτυξη κλπ. Ο μηχανισμός που προτείνουμε είναι ευέλικτος εφαρμόζεται κατά περίπτωση. Λαμβάνονται υπόψη καταστάσεις επιτόπου, οι σχέσεις μας με την τρίτη χώρα και πρόκειται και για σταδιακή προσέγγιση. Μπορεί δηλαδή να εφαρμοστεί σε ένα βαθμό, ίσως ε, όχι σε ολόκληρο τον ε, πληθυσμό της τρίτης χώρας. Πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες κοινοποίηση που δίνουν οι χώρες μέλη, που έχουν συνεργασία με την τρίτη χώρα και πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια ισορροπημένη προσέγγιση και ένα μηχανισμό που εύκολα τίθεται σε εφαρμογή. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση τώρα. Έχει ήδη ξεκινήσει η ψηφιοποίηση για το πις, ήδη γίνεται, αλλά υπάρχει και το αυτοκόλλητο που χρησιμοποιείται. Η ψηφιοποίηση για τις θεωρήσεις είναι για το μέλλον. Θα είναι όντως πιο εύκολο για τους ετούντες, για τα προξενία. Προσπαθούμε και στο τέλος της χρονιάς θα ξεκινήσουμε μελέτη. Η Εστονική Προεδρία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά από αυτού. Και εννοείται ότι θα στήσουμε και τη συμμετοχή και του Κοινοβουλίου και όλων των ενδιαφερομένων στις χώρες μέλη. Πιστεύουμε και εμείς ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η διευκόλυνση ψηφιακή. Για τα τέλη τώρα, το κόστος για τους ανήλικες. Από 0 έως 6 δεν πληρώνουν τίποτα. Από 6 μέχρι 12 ήταν 35 και το κάναμε 40. Κάναμε μια αξιολόγηση τους υπολογισμούς και θεωρούμε ότι πρόκειται για μια λογική αύξηση. Και σας είπα ότι από το 2006 δεν έχει υπάρξει καμία αύξηση. Η κυρία Βαλέρο νομίζω το ρώτησε. Πρόκειται για την κάλυψη του διοικητικού κόστους. Και μετά βέβαια μπορεί να εγκρεθεί ή να αρνηθεί. Η δουλειά όμως θα έχει γίνει από το προξενείο έτσι κι αλλιώς. Από το προσωπικό. Γι' αυτό χρειάζεται το κόστος αυτό. Και πιστεύουμε ότι η δουλεια όμω θα εχει γινει απο το προξενειο ετσι κι αλλιώ απο το προσωπικο γι αυτο χρειαζεται το λογική. Και πιο χαμηλό το κόστος είναι από ό,τι ισχύει στην Αυστραλία ή αλλού. Για την προθεσμία τώρα. Ο κύριος Ντεπρέ γιατί να μην είναι πέντε μέρες. Εμείς πιστεύουμε ότι δέκα μέρες είναι κάτι λογικό πρέπει να γίνουν έλεγχοι ασφάλειας, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτούμε άλλες χώρες, μέλη. Εντάξει, άμα θέλετε το συζητάμε στις διαπραγματεύσει, αλλά με τις αξιολογήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα από το Σέγγεν και τα λοιπά, πιστεύουμε ότι η προθεσμία αυτή είναι λογική για τα προξενία. Τώρα, δακτυλικά αποτυπώματα που θα παίρνει κάποιος εξωτερικός παράγοντας δεν αλλάζουν οι κανόνες. Αυτό ισχύει τώρα το προξενείο είναι αυτό το οποίο αποφασίζει. Πάντα είναι το προξενείο το οποίο αποφασίζει αν θα ε, ανατεθεί σε εξωτερικό πάροχο ή όχι. Δακτυλικά αποτυπώματα κλπ. Και μετά είναι το προξενείο το οποίο έχει το τελευταίο λόγο για το αν θα δοθεί η θεώρηση ή όχι. Οι χώρες μέλη έτσι καλλιώς πρέπει να ελέγχουν τους εξωτερικούς παρόχους. Αυτό υπάρχει ήδη στη ρύθμιση και θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι έλεγχοι αυτοί στο μέλλον για την προστασία δεδομένων κλπ. Είναι πολύ σημαντικό οι χώρες μέλη να φροντίζουν οι εξωτερικοί πάροχοι να εφαρμόζουν πλήρως τους κανόνες. Τώρα για αυτό που ρώτησε ο κύριος Σκουέλιο. Όντως το θέμα της αλλαγής αυτής πρέπει να το δούμε γενικότερα μαζί με την ανακοίνωση που μας οδηγεί σε νέα πολιτική και υπάρχει όντως και η διαλειτουργική προσέγγιση που είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική για την επεξεργασία και τον έλεγχο των αιτήσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι έτσι κάλυψα τα διάφορα ζητήματα και από εκεί και πέρα ευχαρίστω ό,τι άλλε διευκρινήσει θέλετε όταν έχουμε τις διαπραγματεύσει στον τριμερή διάλογο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, γνωρίζετε πως έχουμε καθυστερήσει ε, για την εξετάση του επόμενου θέματος και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι έχουμε μία ακρόαση για τον κώδικα θεωρήσεων και για τις, ε, να το πω, για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Δεν είναι πολιτική δήλωση αυτή που κάνω. Θα αποφασιστεί πώς ε, θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός, όμως αυτή η ακρόαση θα λάβει χώρα στις 10 Ιουλίου, έτσι ώστε να εμβαθύνουμε στις ε, λεπτομέρειες, ε, διότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ε, όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Ε, κύριε εισηγητή, θα θέλατε να πείτε κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσετε. Όχι, όχι μόνο ότι ε, ανυπομονώ να συνεχίσουμε και επιμένω. Ας συνεργαστούμε, ας ε, κάνουμε τη δουλειά έτσι ώστε να κινηθούν τα πράγματα. Φυσικά και έχουμε διαφορές ε, μεταξύ μας οι πολιτικές ομάδες, όμως ας προσπαθήσουμε να επιφέρουμε μια ισορροπία. Και να συνδυάσουμε όλα τα καλά στοιχεία, να συμβιβαστούμε για να περάσει αυτή η νομοθεσία. Και μην ξεχνάτε ότι κάποτε υπήρχαν διάφορα ε, διάφοροι θεσμοί που ήταν ε, των κρατών μελών, ε, κυρίαρχων κρατών μελών. Όμως τώρα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειαζόμαστε μια εναρμονισμένη διαδικασία για την πολιτική θεωρήσεων, παρομοίως και με το άσυλο και με διάφορα άλλα θέματα. Εδώ όμως έχει έρθει η ώρα να κάνουμε επιτέλους δουλειά και να μην επιτρέψουμε να λήξει η θητεία μας χωρίς αποτέλεσμα. Να μην φύγουμε μάδια χέρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να σας πω ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ. Σας ευχαριστώ πολύ στις 27 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί το σχέδιο έκθεσης και σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το 27, μια ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Τάνια Φαγιόν στην οποία θα δώσω αμέσως το λόγο έτσι ώστε να παρουσιάσει το θέμα αυτό χωρίς καμία καθυστέρηση, ακριβώς διότι έχουμε καθυστερήσει. Τάνια λοιπόν έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει τις ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Και εδώ πρόκειται για πολύ δύσκολο θέμα, δύσκολο νομοθετικό έργο. Νομίζω πως ε, είναι μεταδοτική αυτή η δυσκολία. Αν θυμάστε καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τους κανόνες για τους, ε, την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα το 2017 και μετά από μια περίοδο ε, συνεχόμενων έντονων εσωτερικών ελέγχων στα, σε έξι κράτη-μέλη του Σέγγεν έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Νορβηγία και η Σουηδία συνεχίζουν να διεξάγουν ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα, έχοντας ξεπεράσει τη μέγιστη περίοδο που είναι τα δύο χρόνια. Οι λόγοι είναι οι συνεχιζόμενες ε, δευτερογενείς μετακινήσεις. Εμείς ζητούμε να καταργηθούν οι εσωτερικοί ελεγχοί και να αποκατασταθεί η ζώνη του Σέγγεν αμέ, αμέσως. Οι έλεγχοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι παράνομοι. Και εδώ πρέπει να ληφθούν αυτά τα στοιχεία υπόψη. Στην πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή νομίζω πως ε, όπως πιστεύουν και όλοι οι συνάδελφοι, θεωρείται ότι προσπαθούμε να νομιμοποιήσουμε παράνομες πρακτικές. Στις 25 Απριλίου συζητήθηκε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας και μετά υποβλήθηκαν πάρα πολλές τροπολογίες, πολλές από αυτές ε, παρόμοιες. Δεν θα είναι λοιπόν δύσκολο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που πηγαίνουν στην τελείως αντίθετη κατεύθυνση ε, και θα είναι δύσκολο να βρούμε κοινά στοιχεία όμως ο κύριος στόχος ε, δικός μου παραμένει να ε, χαρακτηριστούν παράνομοι και αδικαιολόγητοι οι ελέγχοι στα εσωτερικά σύνορα και να καταργηθούν. Θέλω λοιπόν να σας ε, ρωτήσω, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζώνη του Σέγγεν. Η απάντηση είναι θετική, είναι ναι. Μπορούμε επομένως να συμφωνήσουμε ότι οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν δεν μένει άλλη επιλογή. Χρειάζεται λοιπόν να συζητηθούν οι προποθέσει να υπάρχουν μεγαλύτερε ε, ασφαλιστικές δικλίδες. Η έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα ούτε είναι τόσο σημαντικοί, ούτε και προσφέρουν κάτι και πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα χρονικά όρια, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Η γραμματεία μας έστειλε την πρώτη εκδοχή των ε, τροπολογιών χθε. και με τους σκιώδεις εισηγητές θα συζητήσουμε την προσέγγιση μου, η οποία κιόλας ε, περιγράφεται στο σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα λοιπόν να λάβω την ευκαιρία για να πω δύο λόγια γενικιά, γενικότερα ε, για την κατάσταση στη ζώνη του Σέγγεν. Νομίζω πως έχει συζητηθεί και πριν ότι η εσωτερική έλεγχοι στα σύνορα ε, λάμβαναν χώρα ακριβώς για να ε, προλαμβάνουν δευτερογενείς μετακινήσεις ε, και αυτό ε, είναι κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση στη Γερμανία. Ε, ο, το Υπουργείο Εσωτερικών άρχισε να απορρίπτει αιτήσει ασύλου και επέβαλε ε, πλήρης ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα. Αυτό έχει μόνο είναι παράνομο, αλλά θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του Σέγγεν. Πολύ φοβάμαι ότι η συνέχεια θα είναι συζήτηση για την μεταρρύθμιση του συνολική δέσμης μέτρων για το άσυλο. Ας περιμένουμε όμως να, δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου θα, και θα συζητηθεί το θέμα αυτό στις Βρυξέλλες. Βλέπω ε, όμως ότι το Συμβούλιο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, είναι αδικαιολόγητη αυτή η στάση του και διακυβεύεται το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης. Στην Αυστρία, στα σύνορα με την Σλοβενία, την ε, Δευτέρα που μας έρχεται, θα γίνει μια μεγάλη άσκηση για την προστασία των ε, συνόρων με τη συμμετοχή των, της ειδικής ομάδας Πούμα, ε, μιας ομάδας του Τη ε, το, της με συνεργασία του στρατού και της αστυνομίας. Το ε, υπόθεση της άσκησης είναι πώς να, ε, πώς να επιστρέψουν, να επαναπροωθηθούν ομάδες, μεγάλες ομάδες μεταναστών που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα από την Σλοβενία. Ε, η Σλοβενία έχει επίσης εντοπίσει την ανάγκη για τέτοιες ασκήσεις. Τώρα φαίνεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για το άσυλο, όμως ε, έχει αποτύχει μέχρι τώρα το όλο εγχείρημα και η στάση του Συμβουλίου υπονομεύει οποιαδήποτε έβρεση ευρωπαϊκής λύσης στο πρόβλημα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν θέμα, μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, γι' αυτό λοιπόν ε, έχω μεγάλη περιέργεια να ακούσω την άποψη των σκιωδών εισηγητών. Γνωρίζω ότι μας στηρίζουν όλοι ε, και θα πρέπει να έρθουμε με ενωμένο μέτωπο απέναντι στο Συμβούλιο και την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Τάνια, είναι όντω μεγάλη πρόκληση για το θέμα αυτό και σίγουρα πρέπει να αναφερθούμε και στο γενικότερο πλαίσιο Δυστυχώς λείπουν πολλοί σκιώδες εισηγητές, εκτός από την Ποντήλ. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας δώσω πρώτη το λόγο και στη συνέχεια στους επόμενους συναδέλφου. σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Τάνια, διότι θεωρώ πως ε, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Και να δηλώσω ευθέως ότι στηρίζουμε τις προτάσεις ε, της ε, Τάνια, τις συμβαστικέ ε, τροπολογίες. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να τις στηρίξουμε στο σύνολό τους. Να γυρίσω όμως λίγο πίσω στο χρόνο. Να δούμε το γενικότερο πλαίσιο στην Σουηδία. Εγώ επηρεάζομαι άμεσα από τους ελέγχους που ασκεί η Σουηδία στα σύνορα. Στην ε, νότια Σουηδία που μένει η μητέρα μου για να περάσω πρέπει να πάρω το τρένο και εκεί υποβάλλομαι σε ελέγχους. Οι έλεγχοι στα σύνορα αρχικά ήταν πάρα πολύ σκληρή. Ήδη από τη Δανία κοιτούσαν τα διαβατήρια, σε έλεγχη αστυνομία. Ε, τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουμε επιστρέψει σε περιστασιακούς ελέγχους, αλλά από τη σουηδική πλευρά. Το σκεπτικό πίσω από αυτούς τους ελέγχους είναι να μείνουν έξω οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες. Στην ουσία όμως, όταν φτάνει στη Σουηδία, δεν έχει νόημα να ασκείς ελέγχους, διότι αν θέλει κάποιος θα φτάσει. Ε, στη Σουηδία βέβαια επικαλούνται τη δημόσια τάξη για τους ελέγχους και τα λοιπά, όμως δεν θεωρώ ότι αυτοί οι έλεγχοι εξυπηρετούν κάποιον ουσιαστικό σκοπό και δεν ε, πιστεύω πως πρέπει να ε, χορηγήσουμε άδεια για να ε, δοθεί παράταση σε αυτούς τους ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, πώς θα πρέπει να αντιθράσουμε θα μου πείτε, θα πρέπει να δεχτούμε μια επιδείνωση της κατάστασης μόνο και μόνο επειδή τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις ε, προκλήσεις. Το θέμα νομίζω εδώ, το ζητούμενο είναι η εναρμόνιση. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε επιδείνωση της εναρμόνισης, πισωχυρίσματα, ιδιαίτερα στη μεταναστευτική πολιτική. Βλέπουμε ότι επιδεινώνεται η κατάσταση μέρα με τη μέρα. Και οι κανόνες που έχουμε νομίζω πως χάνουν σε ισχύ και χάνεται ε, και η προσοχή της ε, κοινή γνώμης. Θα πάμε στις ε, συναντήσεις όμως των εισηγητών και θα συζητήσουμε το θέμα με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ναι, φυσικά θα συζητήσουμε το τι συμβαίνει και θα μας ενημερώσει και η Προεδρία στο τέλος. Η Ναταλή όμως έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Κλωτ. Η Σοφίν Φελτ δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί έπρεπε να εξετάσει κάτι φακέλους. Ευχαριστεί βέβαια την ε, Τάνια Φαγιόν και λέει πως πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για την ενότητα, για τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ε, ομάδα μας ε, συμφωνούμε με τη δουλειά της Τάνια. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό πάντως για τη συνέχεια θα δούμε στην ομάδα μας αν θα υπάρχει η αναγκαία ευελιξία ώστε να αποφύγουμε όσο γίνεται περισσότερο κατακαιρματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνοχή είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ. Η Σοφή θα μιλήσει με την Τάνια σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ναταλή, ναι, πολύ λογικό αυτό που λες. Τώρα Ευρω... το Συμβούλιο να μιλήσει, να μας πει τι κάνει το Συμβούλιο από αυτού. Κύριο Σέκοφ, εκ μέρους της Προεδρίας, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να έρθω και να σας μιλήσω εκ μέρους του Συμβουλίου τώρα που είμαστε στις τελευταίες μέρες ουσιαστικά της Βουλγαρικής Προεδρίας. Πρέπει να παραδεχτώ ότι οι τελευταίοι έξι μήνες δεν ήταν μια εύκολη περίοδος, όχι μόνο για μας, ούτε και για τις άλλες χώρες μέλη στο Συμβούλιο και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τον ε, κώδικα Σέγγεν, να ξέρετε ότι εμείς κάναμε τη δουλειά μας και χαίρομαι που μπορώ να σας ενημερώσω ότι το Συμβούλιο πέτυχε το στόχο που φαινόταν να ήταν mission impossible πριν από λίγους μήνες. Στις 19 Ιουνίου λοιπόν οι Ευρωπαίοι πρέσβοι ενέκριναν ανατολή εκ μέρους του Συμβουλίου για διαπραγματεύσεις όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού για τους ελέγχους ε, στα σύνορα που εισήχθη προσωρινά για ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Βάσει της εντολής αυτής λοιπόν, η επερχόμενη Αυστριακή Προεδρία θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άπαξ και έχει οθετηθεί η θέση. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο χώρος Σέγγεν έχει προσφέρει πολλά ωφέλη στους Ευρωπαίους. Η συμφωνία στο Συμβούλιο θέλει ακριβώς να διατηρηθούν αυτά τα ωφέλη και αυτά τα επιτεύγματα. Η προτινόμενη τροποποίηση θα επιτρέψει στις χώρες μέλη να επανισάγουν εσωτερικούς ελέγχους για τους ίδιους λόγους για μια συνολική περίοδο το πολύ ενός έτους. Θα περιλαμβάνει βέβαια και διάφορες ρήτρε ασφαλείας που θα πρέπει να ισχύουν για να ε, τηρηθεί η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των μέτρων αυτών. Να υπάρχει αξιολόγηση κινδύνου, ε, διαβούλευση λοιπά. Όταν ο έλεγχος στα σύνορα γίνεται για πάνω από 6 μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γνωμοδοτεί. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και πάλι για την πρόσκλησή σας και ευχαριστώ και για την προσοχή σας που με ακούσατε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη δουλειά σας, Προεδρία. Τάνια, εντάξει, οι σκιώδες εισηγητές θα πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Θέλεις να απαντήσεις και μετά να συνεχίσουμε. Ναι, ευχαριστώ, Κλόντο. Σύντομα θέλω να απαντήσω στο Συμβούλιο. Ε, σημειώνω τη θέση των ε, συνεισηγητών εννοείται ότι διαβάζω πολύ προσεκτικά το κείμενο του Συμβουλίου. Αυτό που βλέπω και μπορώ να πω τώρα είναι ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία στην εντολή του Συμβουλίου. Λυπούμε όμως που δεν απαιτείται η συμμετοχή του Συμβουλίου για την υπερεισαγωγή των ελέγχων τον πρώτο χρόνο. Αυτό θυμίζει αυτό που προτείνω εγώ στην εκθεσή μου. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να παίξει πραγματικά το ρόλο του θεματοφύλακα των συνθήκων και να αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση που ο δεν τηρείται. Και πρέπει να δούμε ότι η Επιτροπή έχει γίνει πολύ πολιτική, γιατί μερικές φορές δεν αντιδράει, παρόλο που ξεκάθαρα κάποιες χώρες μέλη παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει στις διαπραγματεύσεις. Όπως λέτε και εσείς, πολύ ευαίσθητο ζήτημα αλλά νομίζω ότι οι συγκητές θα ανταπεξέλθουν με υπευθυνότητα. Ευχαριστώ, Τάνια, που είπες και αυτό ότι η Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων, όντω. Η Επιτροπή θέλει να αντιδράσει σε αυτά. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να παρέμβω αρχικά, αλλά ε, εντάξει, μπορεί να μην ε, θέλετε, αλλά σέγγεν αυτό. Ναι, κοιτάξτε, εμεί συμφωνούμε με το σημείο κίνηση τη εισηγήτρια. Ότι δηλαδή πρέπει να διατηρήσουμε το Σέγγεν. Το θέμα είναι πώ θα το πετύχουμε αυτό καλύτερα. Και με την πρότασή μα, όπω εξήγησε έτσι τον Απρίλιο, δεν προσπαθούμε να καταργήσουμε το σύστημα προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τις ρήτρες ασφαλείας όσον αφορά τον κώδικα για τα σύνορα, ώστε να τα αποκρίνονται καλύτερα στις σημερινέ προκλήσεις. Υπάρχουν οι ανώτατοι περίοδοι στον κώδικα σύνορων Σέγγεν από το 2013 μόνο. Και όσον αφορά την διακυβέρνηση του Σέγγεν, γι' αυτό έχουν μπει, αλλά συμφωνήθηκαν σε άλλα πλαίσια για πιο μακροχρόνιες απειλές στην ασφάλεια που δεν υπήρχαν τότε έτσι όπως υπάρχουν σήμερα. Οπότε προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το μηχανισμό Σέγγεν για να ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτές τις απειλές. Βέβαια υπάρχει και συζήτηση για την ανώτατη περίοδο που θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε για τους εσωτερικούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Αλλά ρήτρες ασφαλείας θα πρέπει να υπάρχουν με συνεργασία και με τη συμμετοχή και των χωρών που έχουν επανεισάγει τους ελέγχους στα σύνορά τους. Ο τριμερής διάλογος λοιπόν θα επικεντρωθεί προφανώς σε αυτό, στις ρήτρε ασφαλείας υπάρχει το θέμα του ρόλου του Συμβουλίου ή όχι εφόσον υπάρξει μακροχρόνια παράταση για την, τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Είναι ο Πρόεδρος. Ωραία. Όλοι θα είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στον τριμερή διάλογο. Δεν ήθελα να ξέρω και τη γνώμη σας για αυτά που είπε το Συμβούλιο, αλλά εντάξει, θα μας τα πείτε κάποια άλλη φορά. Ωραία, Τάνη. ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνω τη συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί έχουμε θα συνεχίσουμε φυσικά κάποια άλλη στιγμή τη συζήτηση και στους τριμερείς διαλόγους. Ωραία. Um, Συνάδελφοι, επόμενο μας θέμα είναι η κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Γυναικών για το εμπόριο γυναικών και παιδιών ε, στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Ε, παρακαλώ να μας δώσετε δύο λεπτά να οργανωθούμε. And this scheduled for Για τις 10.30 είναι προγραμματισμένη αυτή η ακρόαση. 10.30. Thanks.